Να σας πληροφορήσω ότι βάσει του άρθρου 231 παράγραφος 4 του κανονισμού δεν υπήρξε καμία αίτηση για ψηφοφορία στο διορθωτικό το οποίο αναφέρθηκε. Ανακοινώθηκε χθε στις 5 η ώρα, επομένως το διορθωτικό αυτό θεωρείται εγκεκριμένο.